Madame la Présidente, je vais ouvrir la séance et après je vous. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα σας δώσω το λόγο. Θέλετε για κάτι στη Ωραία. Καλημέρα λοιπόν. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχω μία ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες σας υποβάλλω.